La séance est ouverte. Άρχεται η συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι. Λέτε ησυχία παρακαλώ. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας και προτείνω να ασχοληθούμε με τα σημεία 6 και 7 ανταλλαγή απόψεων για τις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού του 2014. Ξεκινήσαμε δίμηνη καθυστέρηση το χρονοδιάγραμμα, γιατί χρειάστηκε χρόνος για να οριστικοποιηθεί η πολιτική συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το 2014 είναι η πρώτη χρονιά του πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι πριν από δύο εβδομάδες μας παρουσίασε το σχέδιο του προϋπολογισμού, την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνήσαμε με τη Λιθουανική Προεδρία και δεδομένης αυτής της καθυστέρησης στην έναρξη των εργασιών να οργανώσουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο 2 με 3 Σεπτεμβρίου. Στη συνεδρίαση των συντονιστών πριν από λίγο εγκρίναμε τους πολιτικούς προσανατολισμούς για την εντολή που θα αναθέσουμε προς την ε, εισηγήτριά μας την Αν για τον πρώτο τριμερή διάλογο και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γένσεν για να μας κάνει μια σύνοψη της κατάστασης την οποία θα συμπληρώσει η κυρία Αχνέ, εισηγήτρια για τα για όλα τα τμήματα. Αν Γένσεν πρώτα και μετά η κυρία Χολμάια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την ε, το σχέδιο της σύστασης, το σχέδιο της εντολής ε, για τον τριμερή διάλογο που την συνομολογήσαμε με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες τριμερής διάλογος δεν θα γίνει τον Ιούλιο εξαιτία καθυστέρηση ε, της υποβολής του σχεδίου προπολογισμού, αλλά θα γίνει στι αρχέ Σεπτεμβρίου αυτή τη φορά. Έχουμε καταρχήν την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη τη θέση του Συμβουλίου. Θα συμπληρωθεί λοιπόν το κείμενο όταν υποβληθεί και η ανάγνωση, το αποτέλεσμα της ανάγνωσης από το Συμβούλιο. Το σχέδιο σύστασης είναι αρκετά σύντομο. Περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, που είναι πολύ σφιχτό. Και επίσης αναφέρεται και στο στην κατάσταση που δημιουργήθηκε με τις πληρωμές. Και εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα, σφιγμένα και θα συνεχίσει το θέμα των πληρωμών να εξετάζεται στις διαπραγματεύσεις. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για έναν προϋπολογισμό θύνοντα. Μείωση κατά 6% στις αναλήψεις υποχρεώσεων και 5,8% μείωση στις πιστώσεις πληρωμών. Οπότε ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συρρυκνώνεται. Για τους τίτλους τώρα, τα διάφορα κεφάλαια του προϋπολογισμού, το σχέδιο σύστασης σχολιάζεται τα ποσά. Αυτό που δεν κατανοήσαμε είναι ότι γιατί το κονδύλιο για την έρευνα, το πρόγραμμα COSME, και το αέρασμος, θέμα δηλαδή ανάπτυξης δεν εφοδιάζονται με αρκετά κονδύλια τουλάχιστον σε επίπεδο front loading για το 1β το κεφάλαιο 1β την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι, είναι πολύ σημαντικό θέμα Και εκεί έχουμε ένα front loading για ένα διετές πρόγραμμα και στη συνέχεια θα συνεχίσει το πρόγραμμα ή θα χρηματοδοτηθεί από κοινωνικό ταμείο, που σημαίνει ότι θα μειωθούν άλλα προγράμματα για το 2014. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αργότερα με τη χρηματοδότηση. σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ηθαγένεια. Για τα προγράμματα της ηθαγένειας είχαμε σημαντικές περικοπές. 20 με 25%. ενώ έχουμε αυξήσεις ε, για τα προγράμματα της Ευρώπης για τους πολίτες και τα δικαιώματα των πολιτών Επίσης, ε, στο τίτλο 4, εξωτερικές υποθέσεις. Και εκεί έχουμε μειώσει σημαντικές. Επίσης, σε θέματα υψηλής προτεραιότητας, αναπτυξιακές πολιτικές, πολιτικές γετνίασης. Εκεί, για την Ούνρα, για παράδειγμα, ε, στη βοήθεια για την Παλαιστίνη, έχουμε δραστική περικοπή του ποσού σε σχέση με τις ε, ανάγκες που προβλέψαμε. Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές δαπάνες, μας προβληματίζει η εκκρεμωδικία στο δικαστήριο και δεν ξέρουμε αν θα χάσει το Συμβούλιο την υπόθεση προσφυγής εις βάρος του που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα θέματα των μισθών. Αν τελικά το δικαστήριο δικαιώσει τους ε, ε, ευρωυπαλλήλους, θα υπάρξει ένα κονδύλι που θα χρειαστεί χρηματοδότηση και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, γιατί είναι πιθανό να χάσει το Συμβούλιο. Και το θέμα των οργανισμών επίσης. Είχαμε το πρωί ακρόαση με μερικούς, ε, κάποιους οργανισμούς που μας εξήγησαν την ανησυχητική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. και το πώς ε, αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ε, μειώσεις που θα γίνουν σε προσωπικό στις υπηρεσίες, στις, στους οργανισμούς δηλαδή. Επίσης, μειώθηκε το κόστος κάποιων οργανισμών για να επιτραπεί σε άλλους οργανισμούς να επεκταθούν. Οπότε κάποιοι οργανισμοί εξαιτίας αυτών των περικοπών δεν θα μπορέσουν καν να ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Επίσης, οι ε, ειδικέ επιτροπές ε, θα εξετάσουν τους τομείς ενδιαφέροντός τους και θα υποβάλουν γνωμοδοτήσεις. Ήδη πολλές επιτροπές έχουν συντάξει γνωμοδοτήσεις για τους συγκεκριμένους τομείς που είναι αρμοδιότητά τους. Τέλος, πιλωτικά προγράμματα και παρασκευαστικές δράσεις. που εμπίπτουν στον γενικό προϋπολογισμό για το 2014. Η διαδικασία που ισχύει προβλέπει την υποβολή των προτάσεων, σχεδίων και προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στη συνέχεια εκτιμά κατά πόσο είναι εφικτές αυτές οι προτάσεις. 162 προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτά 132 αφορούσαν νέες προτάσεις και 30 ήδη υπάρχοντα προγράμματα. οριστικός κατάλογος των προγραμμάτων που, είναι, αφορούν 174,15 εκατομμύρια υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό που έχουμε διαθέσιμο, που είναι 50 εκατομμύρια για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και 40 εκατομμύρια για τα πιλωτικά προγράμματα. Βέβαια έχει κάνει και αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 28 προγράμματα έχουν ε, βαθμοδολογηθεί με άριστα, ε, θα χρηματοδοτηθούν. Ε, μετά είχαμε β, μερικά προγράμματα που είναι εφικτά αλλά θα χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τρέχοντα προγράμματα ή θα κρυθούν ανέφικτα. Τις πληροφορίες αυτές θα σας τις στείλουμε με λεπτομέρειες. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για να αποφασίσουμε ποιες προπαρασκευαστικές δράσεις και προγράμματα θα, θα προωθήσουμε και ποιες όχι. το συνολικό ποσό που ίσως χρειαστεί για τα προγράμματα αυτά και τις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις είναι ένα πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα είναι τα ανώτατα όρια στις διάφορες κατηγορίες. Και αυτά τα κατόφλια, τα ανώτατα όρια θα μας περιορίσουμε. Είναι σαν να προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Στην προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο... γίνεται και όσο πολλε, πιο πολλές προτεραιότητες να υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να βρούμε και εφικτά προγράμματα και προγράμματα που θα είναι και αποτελεσματικά και θα επιτύχουν. Αυτά για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Από την πρώτη συνάντηση που είχαμε τις επιτροπές μετά την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού από τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι είναι κυρίως ανησυχία. Γιατί με το νέο πλαίσιο έχουμε χαμηλότερα ποσά, μικρότερα ποσά και κάποια σχέδια έρευνας. Ξεκινούμε με κάποια μείωση σχεδόν 13% και τα επόμενα χρόνια έχουμε σταδιακή αύξηση. Αλλά είναι παράδοξο Απ' τη μια να μιλάμε για την ανάγκη ανάπτυξης ε, και απ' την άλλη να μειώνουμε τα κονδύλια για την έρευνα. Πάντως, επαναλαμβάνω, η πρώτη μου εντύπωση από τη συνάντηση που είχα με τις αρμόδιες επιτροπές είναι απογοήτευση και ανησυχία για την κατάσταση. Δεν αναμένονται και πολύ εύκολες διαπραγματεύσεις δηλαδή. Ευχαριστώ, Άννα. Για λίγη αισιοδοξία η κυρία Χολμαϊά. Κυρία Πρόεδρε, χαμογέλασα όταν είπε η κυρία Γέντσεν ότι θα πρόκειται να είναι δύσκολε οι ε, διαπραγματεύσει. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Και νομίζω ότι έχετε αφήσει τα ίχνη σα ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό και νομίζω ότι και πάλι θα πρέπει να ακολουθήσουμε πιο αυστηρή προσέγγιση. Να σα μιλήσω για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Όπως αναφέραμε και την προηγούμενη φορά και στην προ... προπροηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, ε, τότε δεν είχαμε ακόμα λάβει τις τροποποιήσεις του καταστατικού για το προσωπικό, ούτε και τις τροποποιήσεις του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Όντως, ε, δύο έτη πάγωμα το 2013 και το 2014 του μισθού και αυτό μειώνει όντω τον προϋπολογισμό κατά 0,82% και άρα παρουσιάζεται σαφής ε, μείωση κοιτώντας ε, τι έγινε και τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες ε, στα τέλη της θητείας με τις συνέπειες που συνεπάγεται το τέλος αυτό της περίοδου μιλάμε όχι για 2,2 αλλά για 2,15. Μιλάμε όμως για το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης γιατί είναι, ξέρετε, πολύ ακριβή περίοδος αυτή η τελική περίοδος. Αύξηση 0,76% ε, και προσθέτοντας λοιπόν αυτά τα δύο και υπολογίζοντας ε, το σύνολο έχουμε 2,47% αύξηση και αναφερέσουμε την Κροατία είμαστε στο μείον 0,44% άρα συνολικά βρισκόμαστε σε αρνητικό πρόσημο αν ληφθούν υπόψη όλα και ο πληθωρισμός. Και γενικά να πω ότι πριν την πρώτη ανάγνωση και πριν την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα δούμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ε, Επιτροπή των Περιφερειών και την ΕΟΚΕ, όπου υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία, από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία και άρα θα πρέπει να αλλάξουν τα αριθμητικά στοιχεία, αν μεταφερθεί ένα <coughs> κομμάτι στο Κοινοβούλιο των Επιτροπών αυτών και θα πρέπει να λάβουμε εμείς ένα κομμάτι λοιπόν αυτό και έτσι αυτές οι θέσεις δεν θα προκύπτουν πλέον, δεν θα ανακύπτουν στον προπολογισμό των δύο επιτροπών. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε καταρχάς την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Να δούμε αν ε, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις ε, στο Κοινοβούλιο. Και να δούμε ασφαλώς το Σεπτέμβριο τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Αλλά γενικές ε, γραμμές μιλάμε όχι για αύξηση 3,29 αλλά 2,47% στα άλλα θεσμικά όργανα, τα πράγματα είναι ως εξή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέλει αύξηση 0,2% μετά από συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά κάποιες θέσεις προσωπικού και συμφώνησαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για το 0,2% αυτό. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θέλει μείον 3,2% βάσει διάφορων παραγόντων που έχουν να κάνουν με το ελεγκτικό συνέδριο το ίδιο. Η ΕΟΚΕ θέλει αύξηση 0,7% η Επιτροπή των Περιφερειών 2,2%. Ο διαμεσολαβητής μεγαλύτερη αύξηση 3,8% και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων 10,1%. Και συμπεριλαμβάνω και τις συζητήσεις ε, και να σας πω ότι ο προϋπολογισμός για την προστασία του, των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ περιορασμένος και άρα κάποιες προσαρμογές δεν μπορούν να γίνουν σε μία νύχτα. Θα πρέπει να γίνουν στη διάρκεια των επομενων δυο 2-3 ετών και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συν 3,2% για τα υποχρεωτικά μέτρα αλλά και για τα μέτρα ασφάλειας. Αλλά και λαμβάνοντα υπόψη την αυξανόμενη τιμή των ενοικίων αν ε, το περασμένο ήτος λοιπόν ε, το ενίκιο ήταν για τρεις μήνες και τώρα ε, μιλάμε για μια δωδεκάμινη περίοδο, ναι, ομολογουμένως ο προϋπολογισμός είναι πιο υψηλός, αλλά δεν σημαίνει ότι ξοδεύονται παραπάνω χρήματα. Αυτά λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία στα άλλα θεσμικά όργανα δεν υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα και στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει διαφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Γένσεν για το έργο της και την προεργασία αυτή που έγινε για την εντολή και για τον τριμερή διάλογο και την ευχαριστώ θερμά γιατί επέτρεψε τη συμμετοχή και των ε, πολιτικών ομάδων και τη συμβολή τους, τη συνεισφορά τους. Ως προς τα σχόλια δεν έχω και πολλά να προσθέσω, συμφωνώ με τους προσανατολισμούς. Πάντως για τη δημοσιονομική διαδικασία του 2014 έχουμε πολλούς αγνώστους χι ακόμη. Ο χρόνος προχωρά, αλλά τα θέματα αυτά δεν έχουν διαλευκανθεί. Υπάρχει ένα μια προκαταρκτική συμφωνία του δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από την προκαταρκτική αυτή συμφωνία ε, απορρέουν πολλές αλλαγές για τους προϋπολογισμούς. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περισσότερες πληροφορίες για το πότε θα υποβάλει το διορθωτικό της προϋπολογισμό, το διορθω επιστολή για τη διόρθωση της πρότασης του προσχεδίου προϋπολογισμού, γιατί μιλήσαμε για την εγγύηση για τους νέους ε, και την μεταφορά κονδυλίων εκεί. Οπότε και μόνο αυτό θα τροποποιήσει την πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2014. Και για την, προκαταβολή, για την προκαταβολή αυτή θα πρέπει να βρούμε μια, ένα αντιστάθμισμα μειώνοντας άλλα ποσά, ίσως τη διευκόλυνση του Connecting Europe το συνδέοντας την Ευρώπη. Πολλές αλλαγές ήδη προβλέπονται και δεν ξέρω πώς θα εργαστούμε και φυσικά όλα εξαρτώνται και από την ανάγνωση του Συμβούλιο. Αλλά αν δεν ε, λάβουμε και την νέα πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς με τι βάση θα εργαστούμε και πού θα προτείνουμε τροπολογίες. Ό,τι αφορά το backloading, την επιστοβαρή χρηματοδότηση για κάποια προγράμματα, πώς θα επηρεαστούν τα προγράμματα από το backloading για το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη και για άλλα προγράμματα. Είχαν προβλεφθεί κάποια κονδύλια για τα πρώτα χρόνια. Τώρα λέμε ότι μερικά από τα κονδύλια αυτά θα περάσουν σε backloading. Ήδη έχει πληγεί το συνδέοντας στην Ευρώπη από την Συμφωνία για το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και έχει περικοπεί αρκετά. Πώς θα επηρεαστεί η εφαρμογή και του Connecting Europe Facility και άλλων προγραμμάτων από τις περικοπές. Για τους οργανισμούς επίσης θα έχουμε, με τους οργανισμούς θα έχουμε πρόβλημα. Το συζητήσαμε και το πρωί. Γιατί έχουμε επέκταση της εντολής πολλών οργανισμών και αύξηση των αρμοδιοτήτων τους και ταυτόχρονη μείωση των προϋπολογισμών τους. Και αν δεν κάνω λάθος, το Συμβούλιο κάνει μια ενδελεχή ανάλυση των οργανισμών και επικεντρώνει τις περικοπές που προτείνει στους οργανισμούς. Οπότε θα επιδεινωθεί το πρόβλημα με την ανάγνωση του Συμβουλίου για τους οργανισμούς. Σε ό,τι αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα... θα υποβληθούν άλλων τροπολογίες και από τις ε, άλλες επιτροπές. Οπότε θα χρειαστεί να λάβουμε μια πολύ δύσκολη απόφαση εμείς παίξουμε τους κακούς της ταινία. Ένας ρόλος που δεν με ευχαριστεί καθόλου. Κάθε ευρώ που θα αφιερώνουμε σε προπαρασκευαστική δράση, σε πιλωτικό πρόγραμμα ή στην αύξηση οποιοδήποτε τμήματος του προπολογισμού που κρίνουμε ως προτεραιότητα, θα πρέπει να το αφαιρούμε από το περιθώριο που υποτίθεται θα έχει προβλεφθεί για να, προγραμματίσει την εγγύηση για το νέο το 2016. Αυτό προβλέπει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ό,τι περισσέψει το 2014, 2015, 2016 και 2017 ε, θα χρησιμοποιηθεί για την εγγύηση για τους νέους. Οπότε είναι σαν να μας ζητά κανείς να επιλέξουμε ποιον αγαπάμε περισσότερο, το πατέρα μας ή τη μητέρα μας. Όλα προτεραιότητες είναι. Δύσκολες θα είναι οι επιλογές. Και τελευταία ερώτηση προς την Επιτροπή. αν δεν κάνω λάθος, 0,2 ήταν ε, το περιθώριο πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού, δηλαδή μηδενικό ουσιαστικά. Άρα δεν υπάρχει κανένα απόθεμα ε, για τα απρόβλεπτα ή για ε, απλήρωτους λογαριασμούς. Ούτε καν υπάρχει περιθώριο για προσαρμογές στο κεφάλαιο 5. Αν ε, η απόφαση του δικαστηρίου δικαιώσει τους υπαλλήλους, ε, δεν έχουμε καν απόθεμα για να διορθώσουμε τις μειώσεις που έγιναν προηγουμένως, για να συμπληρώσουμε τους μισθούς. Δεν ξέρω, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για κάθε δεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ο Ντομινίκ Ρικέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Γκαρδιά Ζαμπάλ και με τα οποία συμφωνώ. Την ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που μπόρεσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες να μπορέσουν να διαμορφώσουν την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν σωστή. Να κάνω κάποιες μακρο σκοπικές εισαγωγικά παρατηρήσεις. Το πρώτο που διαπιστώνει κανείς είναι ότι πράγματι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Κάρτια Ζαμπάλ δεν μπορούμε να καλύψουμε το απρόβλεπτο και δεν έχουμε και κανένα τρόπο να προσαρμόσουμε έστω και προς τα κάτω τον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτησίες θα γίνονται ανάμεσα στις διαφορετικές θέσεις του προϋπολογισμού. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση ε, σε αυτό τον προϋπολογισμό ε, ε, που αναφέρεται αν θέλετε στη σύγχρονη αξία του ευρώ μιλάμε για ποσοστά ρευστοποίηση ουσιαστικά. Έχουμε τα ραλ τα οποία εκφράζονται έτσι και αλλιώς μέσα από τον προϋπολογισμό και η μεγάλη πλειοψηφία των πιστώσεων πληρωμών θα στραφούν προς τα αρέστα λικίντε, προς τα ράλ. Τα υπόλοιπα προς ρευστοποίηση. Μετά από κάποιες έτσι περίεργες πολιτικές κινήσεις του Συμβουλίου, προωθούνται υποτίθεται ορισμένες δράσεις και όλοι ανακαλύπτουν ξαφνικά τις χαρές του front-loading και του back-loading. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει σύντομα από ό,τι φαίνεται ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Θα είναι δυνατόν να θέσει ε, στη διάθεση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας κυρίως ένα πρόγραμμα για το σύνολο των προοπτικών που θα μας εξηγήσει το πώς θα λειτουργήσει το front και το backloading καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Γιατί αν αρχίσουμε την μπροστογεμή φόρτιση μετά από διαιτησίες οι οποίες θα είναι ακραίες και στο τέλος θα καταλήξουμε με κάποια κορόιδα ουσιαστικά. Και τα δύο-τρία τελευταία χρόνια κάποιοι θα έχουν πλέον ιτηθεί πλήρως. Όταν λοιπόν το Κοινοβούλιο συμφωνήσει με ένα πολιετές πλαίσιο, το κάνει για το πλαίσιο το οποίο πρέπει να είναι ειλικρινό. Όταν βλέπω την σημασία των προτάσεων που αφορούν το front-loading αλλά και το back-loading, ανησυχώ γιατί αν αυτό είναι κάτι το οποίο διασφαλίζει την ισορροπία της εξαετούς περίοδου. Δεν φαίνεται. Όπως είπα, ο προπολογισμό είναι προϋπολογισμός ρευστοποίησης. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο, καμία νέα δράση και 10% αβεβαιότητα. Είναι, ε, όπως είπα, προϋπολογισμός ρευστοποίησης. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο να διαπραγματευτούμε εδώ συνάδελφοι γιατί δεν υπάρχει τίποτα να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά. Το μόνο στο οποίο πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί είναι το backloading και το frontloading τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά στα πλαίσια των προοπτικών γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε σκληρά για το δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά υπό το άλοθη του ότι, ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ε, θα υπάρξουν δεκάδες ε, ανακατανομές χωρίς να ελέγξουμε εμείς τίποτα. Εδώ θα πούμε ότι η αναδιαπραγμάτευση της αντολής την οποία ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε θα δώσει δυναμική στη δημοσιονομική διαδικασία. Φοβάμαι ότι αυτό θα καταλήξει σε ένα λογαριασμό που θα καλύψει τις ανάγκες των τριών πρώτων ετών και θα οδηγήσει στην διάλυση ορισμένων πολιτικών. Η κυρία Γκουαρδιά Ζαμπάλα αναφέρθηκε σε πολιτικές βασικές για την ανάπτυξη. Είδα πως ξεκίνησαν σε τέτοιου είδους τα πράγματα με τον backloading. Αν πραγματικά πάνε χάλια τα πράγματα σημαίνει ότι μας έχουν σε δουλέψει. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να είναι πάρα πολύ προσεκτική για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμει όλα αυτά κατά τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών. Ευχαριστώ συνάδελφε για την σημαντική παρατήρησή σας. Χάουγκ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα μπορούσα να επαναλάβω όλα όσα είπα σήμερα το πρωί κατά τη συνάντηση με τους οργανισμούς. Αλλά θα περιοριστώ και θα πω το εξής. Αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση για τον προπολογισμό πολύ απλά δεν, μπορέσουν, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Ξέρουμε όλοι πως ε, από τι αποτελείται και πώς ε, καταρτίζεται ο προπολογισμό των οργανισμών. Υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πολιτές Πρόγραμμα, το Πρόγραμμα Εργασίας. Τα προγράμματα που έχουμε εγκρίνει, το έχει κάνει αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε τόσα χρήματα, τόσα κονδύλια. Και τα μεταβιβάζουν αυτά στις ε, ομόλογες ε, γενικές διευθύνσεις, οι οποίες ε, τα πηγαίνουν και αυτές με τη σειρά τους στη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού, η οποία και μειώνει τα ποσά αυτά. Αλλά εκεί δεν σταματάει η ιστορία. Όχι μόνο η εμπειρία μας, αλλά και τώρα η σημερινή πράξη. Τι μας καταδεικνύει, ότι το Συμβούλιο θέλει τα λίγα χρήματα, τα λίγα κονδύλια, τα περιορισμένα κονδύλια τα οποία διατίθενται στους οργανισμούς να περιοριστούν περαιτέρω. στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών ε, μιλήσαμε για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων. Ε, μάλλον δεν μιλήσαμε, αναβάλαμε για το Σεπτέμβριο τη συζήτηση των, της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας ε, για την αυτιλία. Και πολύ απλά δεν υπάρχει κάποια λύση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα δεν μπορεί να πετύχει αυτό που πρέπει να πετύχει με 6,5 εκατομμύρια παραπάνω σε πέντε χρόνια. Είναι αυτό ανοησία πραγματικά. η Επιτροπή Μεταφορών μετά από πρόταση του εισηγητή λέει ότι χρειάζονται όχι 6,5 εκατομμύρια παραπάνω, αλλά 32,5 εκατομμύρια παραπάνω. Τουλάχιστον. Ούτε αυτό το ποσό αρκεί. Πολύ απλά δεν είναι ρεαλιστικά τα ποσά αυτά. Αυτό όμως τι σημαίνει. Ότι η μοναδική δυνατότητα που έχουμε είναι να δηλώσουμε ότι τόσα κονδύλια έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν υπάρχουν παραπάνω, μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Συμβούλιο κάνει και άλλε περικοπέ και δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να πούμε ότι εντάξει δεν θα περιλαμβάνονται πλέον η χ, αρμοδιότητα. Δεν είναι δυνατόν να τα κάνουν όλα. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, να το τελειφθούμε. Δεν είναι δυνατόν να προσθέτουμε καθήκοντα, γιατί όλα είναι ωραία και όμορφα και σημαντικά και τα θέλουμε, αλλά στο τελική ανάλυση αυτά που ως νομοθέτης τα αποφασίσαμε να μην θέλουμε να τα χρηματοδοτήσουμε, να μην θέλουμε να τα πληρώσουμε. Τελεία και παύλα. Είναι οι ίδιοι οργανισμοί. Μόνο στο κοινοβούλιο στέκουν τα πράγματα. Κάτι άλλο επίσης που υπέτυξε και το Μινίκ και το έθεσε και η ΕΝΤΑ. Πότε θα λάβουμε αυτό το amending letter, την τροποποιητική επιστολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την αναφέρει καν για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι αυτό που πρότεινε ως προπολογισμό πολύ απλά δεν είναι εφαρμόσιμο. Θα πρέπει να υπάρχει και μια σχετική κοινοποίηση. Δεν το αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1η, 2η, 3η Ιουλίου η Επιτροπή Προπολογισμών του Κοινοβουλίου συνεδρίασε, του Συμβουλίου συγγνώμη, συνεδρίασε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγήκε και δήλωσε στο κοινό, στη δημοσιότητα, πού θα γίνει front-loading και πού θα γίνει back-loading. Και πού θα γίνει back-loading στον ορίζοντα 2020, στο Εράσμος, άκουσον, άκουσον και πού αλλού. Στην ε, ε, ενέργεια και στις μεταφορές, ασφαλώς. Και πού θα γίνει front loading, επειδή χρειαζόμαστε κατεπηγόντως τα χρήματα εκεί, στο Ίτερ και στον Γαλιλαίο. Μα ποιος πιστεύει ότι τα χρήματα τα οποία έχουν μπει στον loading θα βγουν και θα χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή. Κανείς δεν το πιστεύει και αυτό βγαίνουν και το λένε στο Συμβούλιο και συμφωνούν όλοι υπάλληλοι. Κανένας πολιτικός ηθήνων. Όλοι υπάλληλοι. Πραγματικά είναι για κλάματα. Για κλάματα. Δεν είναι δυνατόν. Και αν δεν έχουμε περιθώρια, το οποίο και αυτό, και γι' αυτό διαμαρτύνονται στο Συμβούλιο και θέλουν ακόμα και στις πιστώσεις να, γίνει, να υπάρχει ένα τέτοιο περιθώριο και γι' αυτό κάνουν περικοπές στις πληρωμές όπου μπορούν προκειμένου να υπάρχουν στις πληρωμές ε, ένα περιθώριο. Μα τι θα γίνει και με το μέσο ευελιξία. Και αυτό το αποφασίσαμε. Μα δεν θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Τι να σας πω, το πράγμα βρωμάει όλο και πιο πολύ. Και βρισκόμαστε εδώ για να διαπραγματευτούμε διάφορες, ε, διάφορα θέματα του προπολογισμού και πλέον δεν μπορώ να καταλάβω πλέον πώς ε, συμπεριφέρεται έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ένωση του Συμβουλίου. Συμβουλίο. Ευχαριστώ κύριε Χάρτονγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σα ε, προκαλέσει εντύπωση το ότι έχω τελείω διαφορετική άποψη από την συνάδελφη Χάουγκ. Να μιλήσω στην συνάδελφο, για τη συνάδελφη Χολμάιερ και να σα πω το εξή. Να ρωτήσω. Έχετε, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αίσθηση κατεπίκοντο σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει για του οργανισμού. Έλαβα ένα σημείωμα ενό δικτύου οργανισμών όπου αναφέρουν ότι οι περικοπές στα κρατη θεωρούν ότι είναι αναγκαιότητα και ότι οι περικοπέ για του οργανισμούς είναι απαράδεκτες. Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ τον λαό και είμαι περήφανο που μπορώ να μιλήσω εκ του λαού μου στην χώρα μου και να πω ότι πραγματικά το βρίσκω ε, απαράδεκτο και δεν το πιστεύω ότι το γράφουν αυτό οι οργανισμοί. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να καταργηθούν οι οργανισμοί. Merci, mon cher collègue, Monsieur Paul Ruby. ευχαριστώ, κύριος Paul ευχαριστώ, Πρόεδρε, και για να είμαστε και πάλι σοβαροί. Νομίζω ότι τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και εδώ πρέπει να συζητηθούν. Χαίρομαι που σήμερα το πρωί συζητήσαμε σοβαρά το θέμα του Εράσμου για τους νέους επιχειρηματίες, γιατί χρειαζόμαστε πολύ απλά ανθρώπους οι οποίοι θα λάβουν την ευθύνη για την απασχόληση και που θα φροντίσουν να σημειωθεί πρόοδο στον τομέα αυτό και είμαι πάρα πολύ περήφανος που σήμερα εδώ ομόφωνα όλες οι ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο δηλώσαμε ότι το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες θα μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο αυτών των προγραμμάτων των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια νέα κουλτούρα που είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας και που υποστηρίζεται άλλωστε και πάρα πολύ έντονα από τους κοινωνικούς εταίρους. Νομίζω ότι για το πρώτο έτος τα 20 εκατομμύρια που προβλέπονται μας δίνουν τη δυνατότητα, ξέρετε, αυτά τα προγράμματα να ανακτήσουμε και την αξιοπιστία μας στα μάτια των πολιτών. Τα καθήκοντα όμως τα οποία ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να παρέμβει εκεί που αποτυγχάνουν τα κράτη-μέλη και μιλάμε και τεράστια αποτυχία των κρατών μελών δυστυχώ σε ό,τι αφορά τα θέματα απασχόλησης. Τα πρόγραμματα λοιπόν αυτά θα πρέπει, που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθήκον μας αυτό. Ε, Τύχη. Έχουμε εδώ τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Ακούσατε τις απορίες των συναδέλφων. Να σας μεθυμίσω ότι η συμφωνία που συνήψαμε στο γραφείο μάλιστα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσία του Ολλανδού Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να αντικατοπτριστούν στους προϋπολογισμούς του 2014 και του 2015, γιατί πέραν του front-loading που ζητούσε το Συμβούλιο, ειδικά για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία για τους νέους και για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είχαμε λοιπόν συμφωνία για το front loading για τις δεύτερες χρονιές στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταξύ του ορίζοντα 2020, του Erasmus Συν και του προγράμματος Κόσμα. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, περιμένουμε την τροποποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2014, ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία. Και μία άλλη ερώτηση είναι ότι στις αποφάσεις που μας ενήγγειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία για τους νέους και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε αμέσως μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στις δηλώσεις που έκανε και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησε για 8 δισεκατομμύρια. Ενώ μέχρι τότε σε όλα τα έγγραφα και στις ε, δηλώσεις που ακούγαμε αναφέρονταν 6 ε, δισεκατομμύρια. Έχουμε σήμερα περισσότερες πληροφορίες για το από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια. Και, και ε, σωστά είπε ο Ντομινίκ Ρικέ, καλές οι προκαταβολές στο front loading αλλά όχι εις βάρος άλλων πιστώσεων που θα καθυστερήσουν. Θα πρέπει η αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σίγουρα και το Συμβούλιο, να έχουν ε, εμπεριστατωμένη και σαφή γνώμη για το τι θα γίνει με τον πίνακα των ανώτατων ορίων για το σύνολο της ε, περίοδου του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου μετά τις αποφάσεις αυτές. Ε, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε αυτά τα σημεία κύριε Γενική Διευθυντά να προσπαθήσω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Ξεκινώντας και οι παρατηρήσεις που έγιναν για το μέγεθος του προϋπολογισμού και την έλλειψη του περιθωρίου. Αυτό είναι μια μηχανιστική αν θέλετε κατάληξη και συνέπεια της κατάστασης την οποία βιώνουμε λίγο πριν το 2014 και του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Οι αριθμοί κατετέθησαν από τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι. Είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση όπου τα ραλ ε, που μένουν είναι σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούν κάποια προγράμματα στα πλαίσια 14-21. Ε, η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της περίοδου αυτής οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι λίγο χαμηλότερες από ό,τι ε, θα φανταζόταν κανείς στα πλαίσια του ενεστώτος του ισχύοντος ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Στην αρχή της επομένης περίοδου το ειδικό βάρος αν θέλετε θα έχει να κάνει με την αποπληρωμή των αποδείξεων του παρελθόντος αυτό δεν είναι περίεργο, αυτή είναι η λογική του συστήματος με το οποίο εργαζόμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μη σας κάνει εντύπωση. Πράγματι λοιπόν και λόγω του ε, σχετικού χαμηλού επίπεδου, χαμηλού ύψους των πληρωμών, κάτι το οποίο μαθηματικά δεν ήταν λογικό ε, να οδηγήσει στην πρόβλεψη ενός διαφορετικού περιθωρίου από αυτό το οποίο προτείνουμε. Τώρα για τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το front loading και το back loading. Εδώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Στο ε, προσχέδιο το οποίο σας έχει πλέον υποβληθεί, δεν είχαμε ενσωματώσει την προσαρμογή η οποία έχει υπάρξει στα προγράμματα τα οποία ήδη αναφερθήκατε, ε, κόσμε ε, Horizon 2020 και έρασμος για όλους. Και θα υπάρξει μια διορθωτική, αν θέλετε, ρύθμιση, ένας διορθωτικός τον μήνα Σεπτέμβριο που θα καλύψει το θέμα αυτό. Τότε θα έχετε λοιπόν τον μήνα Σεπτέμβριο μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι front-loaded και τι είναι back-loaded, για να το πούμε στα αγγλικά, λέει ο τη γαλλική ομιλητής και που αφορούν κυρίως και τα προγράμματα, τις ανάγκες των προγραμμάτων για τους νέους. Τώρα, τα ποσά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην αρχή της περίοδου, στο Α κόσμε Εράσμους για όλους και ορίζον 2020, τα ποσά αυτά δεν χάνονται, δεν θα πάνε χαμένα για το Connecting Europe Facility ή για την ενέργεια. Πρόκειται για ποσά, πρόκειται για πιστώσεις τις οποίες ουσιαστικά σπρώχνουμε για αργότερα που αντικαθιστούν τα ποσά τα οποία είχαν αρχικά προβλεφθεί για τα προγράμματα τα οποία έχουν γίνει ήδη front-loaded και τα προγράμματα, οι πιστώσεις αυτές θα δαπανηθούν, αλλά θα δαπανηθούν σε υστερότερο χρόνο. Γιατί? Το έχουμε εξηγήσει ήδη και θα το επαναλάβω. Το κάναμε γιατί αυτό μας επέτρεπε να καταλήξουμε στην βέλτιστη δυνατή χρήση των πιστώσεων υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Οι εμπειρογνώμονές μας μας εξήγησαν ότι στον τομέα της ενέργειας η θέση σε λειτουργία των προγραμμάτων θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε προβλεφθεί όταν κάναμε εμείς την αρχική πρόταση κατανομής των πιστώσεων. Αντίθετα, για να μπορέσουμε να επανεξισορροπήσουμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων, θα μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε και τη χρήση τους, καλύπτοντας τις προσδοκίες που υπάρχουν στον τομέα της έρευνας, της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων και του Εράσμους για όλους και θα έχουμε στον εύθετο προβλεπόμενο χρόνο τα ποσά που χρειαζόμαστε για την ενέργεια και για τα Connecting Europe. Λοιπόν, Έπρεπε να το διευκρινίσω αυτό για μια ακόμη φορά γιατί είναι σημαντικό. Τώρα για τα υπόλοιπα που ακούστηκαν νομίζω ότι έχω ήδη δώσει κάποιες απαντήσεις. Να πω ότι σε επίπεδο διορθωτικής επιστολής θα υπάρξει η πρώτη, ο πρώτος διορθωτικός ε, προϋπολογισμός ο οποίος θα καλύπτει τις συνέπειες του front-loading. Θα υπάρχει και μια δεύτερη επιστολή ως συνήθως που θα αφορά την γεωργία. Ε, παραδοσιακά γίνεται και θα κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνήθως τα μέσα του μηνός Οκτωβρίου. Λοιπόν αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω μετά από τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Ευχαριστώ. Για τα οκτώ δις για τα 6 ή 8 δις. Τι έχετε να πείτε. Κύριε Πρόεδρε, ξέχασα να απαντήσω σε μία επιπλέον ερώτηση και θα απαντήσω στη δική σας αμέσως μετά. Για τον κύριο Ρικέ, λοιπόν, πράγματι εμείς παράγουμε ένα έγγραφο ε, δημοσιονομικού προγραμματισμού, το οποίο κατατίθεται παράλληλα με τον προϋπολογισμό. Σε αυτό το έγγραφο θα δείτε την περιγραφή των συνεπειών της ανακατανομής των πιστώσεων υποχρεώσεων ε, λόγω του back και front loading. Ε, εκεί κατατίθενται ξεκάθαρα το τι θα γίνει. Τώρα για τα 6 δις ή τα 8 δις. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν κάνει κανένα υπολογισμό. Ο αριθμός τον οποίο εγώ γνωρίζω είναι τα 6 δις. Ε, είναι ο αριθμός ο οποίος έχει συζητηθεί, έχει καθοριστεί αν θέλετε και έχει οδηγήσει στο να καταλήξουμε σε μια πρώτη συμφωνία. Τώρα, αν ε, θέλετε να κάνω λίγο τον Μάντι θα μπορούσα να πω ότι στα πλαίσια των γενικότερων απόψεων αυτών που ανέφεραν αυτό τον αριθμό, τα δύο επιπλέον δις ανταποκρίνονται στο τι θα υπάρξει από το γενικό περιθώριο, το οποίο συνετέθη ε, και θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθούν κάποιες ενέργειες για τη δεύτερη περίοδο. Η ερμηνεία όμως αυτή την οποία μόλις σας έκανα είναι μια πάρα πολύ προσωπική ερμηνεία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας καθησυχάζει ή να μας ανησυχεί η σύμπτωση αυτή των, της αντίληψης της ερμηνείας μας για την τελευταία κατάσταση. Δηλαδή ότι γίνεται μια πολιτική ανακύκλωση των ίδιων αριθμών. Η ίδια αριθμοί, αλλά για διαφορετικές προτεραιότητες από τη μία μέχρι την άλλη σύνοδο κορυφής. Δεν έχουμε σώρευση αριθμών, αλλά τους ίδιους αριθμούς, τα ίδια ποσά που ανακυκλώνονται. Η Μόνικα βιάζεται και πρέπει να μας μιλήσει και για την building policy την πολιτική των ακινήτων. Οπότε ολοκληρώνουμε το θέμα της εντολής ε, για το τριμερή διάλογο και να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Σημείο 27, Μόνικα. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί μιλάμε για δύο κτίρια. Το πρώτο βρίσκεται σε μια δύσκολη ε, περιοχή στην Αγγόλα, αλλά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εκτορικής Δράσης έχει ως πρόθεση να διαμορφώσει με πιο σωστό τρόπο τα πράγματα. Μιλάμε, μιλάμε για έξτρα έξοδα 400.000 ευρώ ανά έτος, αλλά αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου το παλιό κτίριο το οποίο βρίσκεται σε επομένη κατάσταση να με γεννήτρια μέσα σε ένα κτίριο ε, σε γραφεία, σε κτίριο γραφείων ε, προκύπτουν πραγματικά κίνδυνοι για τους υπαλλήλους. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πολλαπλή έκκληση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας η κατάσταση πραγματικά είναι απαράδεκτη για τους υπαλλήλους και γι' αυτό λοιπόν μιλάμε πλέον για ένα νέο κτίριο. Το νέο κτίριο επειδή έχει χτίστη το 2013 και άρα στο σύνολό του είναι φυσικά πιο ακριβό, αλλά πληρεί τις κανονικές προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλου. Επιτέλους δηλαδή, στο μέλλον θα έχουμε 1,46 εκατομμύρια παραπάνω, αλλά θα έχουμε ε, λιγότερο, αν θέλετε, παράπλευρο, μικρότερο παράπλευρο κόστος σε ό,τι αφορά και επίσης 1,127 ε, ε, εκατομμύρια δεν θα τα πληρώσει το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση. άρα συνολικά θεωρούμε ότι είναι σωστή η απόφαση. Άρα θα ήθελα να μην γνωρίζουμε ύστερα μία πληροφορία, Πρόεδρε. Κάναμε πολλές συζητήσεις για τα κτίρια στο Λουξεμβούργο. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό το Δικαστηρίο γιατί εγκατέλειψη το ένα κτίριο και έτσι το Κοινοβούλιο μπόρεσε να συζητήσει με ενοικιαστές και μάλιστα είχαμε και δύο προσφορές και έχουμε έτσι εξοικονομούμε 1,1 εκατομμύρια και έτσι μπορούμε να εξοπλίσουμε το νέο κτίριο με πιο καλές προδιαγραφές και μιλάμε για 5 ε, εκατομμύρια κέρδος σε 25 μήνες. Είναι πολύ θετικό αυτό και ε, επίσης ε, επειδή δεν μιλάμε για επιβάρηση του προπολογισμού, αλλά αντιθέτω για ποσό το οποίο προκύπτει πλανασματικά, δεν χρειάζεται κοινοποίηση και ασφαλώ και αποδεχόμαστε αυτή την αλλαγή. Ε, Σα ευχαριστούμε, κύριε Συγκετριά. Η Συγκετριά μα λοιπόν προτείνει να μην δώσουμε γνωμοδότηση για α, ε, σύσταση αντιπροσωπείας της ΕΙΑΔ στη ΛΟΑΝΤΑ και σας εξήγησε για, για τις δυσκολίες που υπήρχαν και τη σκανδαλώδη κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το κτίριο Γέος στο Λουξεμβούργο, Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για τις οικονομίες που έγιναν χάρη στις προσπάθειές της μεταξύ άλλων. Συμφωνούμε όλοι, πολύ ωραία, οπότε χρειάζεται να ψηφίσουμε για την κτηριακή πολιτική. Μπορούμε όμως να περάσουμε στις υπόλοιπες ψηφοφορίες, σημείο 21. Προγραμματισμός πολιτικής και μακροπρόθεσμες τάσεις. Εισηγητής James Ellis votre euh, voting list. Παρακαλώ, να δούμε τον κατάλογο ψηφοφορία. Έχετε ελπίζω τις κάρτες σας, τις ηλεκτρονικές για την ψηφοφορία. Voilà. Bien. Tout le monde a sa... Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορία Πολύ ωραία. Έκθεση James Ellis. Τροπολογία 2. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο άλλο είναι υπέρ. Κατά. Τρει αποχέ. Ουδή. Εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 3, 4 και 5 του κ. Φεραίρα. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ κυρία Σούζα. Κατά όλοι οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτονται οι τροπολογίες Φεραίρα. Τροπολογία 6. Γκούσταυσον Ματέρα. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Άλτα. Κατά. Πολύ. Αποχές απορρίπτονται. Συμβεβαστική τροπολογία α, κεφαλαίο. Με το συμπεριλαμβανομένη ευρύτερη ερευνητική κοινότητα εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. κτλ. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική Α. Κατά. Τρει κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει η τροπολογία 7 και η τροπολογία της ΑΦΚΟ. Τροπολογία 8 και 9, κάλφιν, μαζί. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ωραία, κατά χάρτων. Αποχές χωρίς αποχές εγκρίνονται. Για τις ιδεολογικές σκέψεις. Τροπολογία Γκούσταυσον Ματέρα. Ο είναι υπέρ. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την γνωμοδότηση της επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξης. Καλά, αν επιμένετε. Έχετε διάθεση για επιπλέον ψηφοφορίε. Ο εισηγητή είναι κατά τη γνωμοδότηση Ρέτζι 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Τέσσερι είναι κατά. Και ο εισηγητή 5. Αποχέ. Μία αποχή. Εγκρίνεται η Ρέτζι 1. Η Ρέτζι 2, 3, 4 και 5 δεν χρειάζεται να ψηφιστούν γιατί είναι εκτός θέματος. 6 και 7 της Ρέγγι μαζί ή όχι. Άντε ξεχωριστά. Ή 6. Ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά. Άλτα. Κατά. Πολύ. Απορρίπτεται. 7 της Ρέγγι. Ποιος είναι υπέρ. Ο εισηγητής είναι επίσης κατά. Και εδώ. Κατά. 6 κατά, αποχές εγκρίνεται και αυτή, η 7 της Ρέγγι. Ρέγγι 8 και 9 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, ο γιατί είναι υπέρ, 8 και 9 ποιος είναι υπέρ, κατά 2 αποχές, μία αποχή, εγκρίνονται. Μας ενδιαφέρει και η γραμματότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Ναι. Ένα και δύο μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Τρεις κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία β κεφαλαίο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τρεις κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. θα γίνει νέα παράγραφος 5α. Οι 3 και 4 της ΑΦΚΟ καλύπτονται από την συμβαστική τροπολογία Β κεφαλαίο. Οι 5 εν μέρη από τη νέα παράγραφο 5. Αλλά μπορούμε να ψηφίσουμε την ΑΦΚΟ 5 ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. 2. Αποχές εγκρίνεται ως προσθήκη. ΑΦΚΟ 6. 7 και α. Προσθήκες. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της ΑΦΚΟ 6. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΑΦΚΟ 7. Ως προσθήκη. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές μία αποχή εγκρίνεται. Αύκο α κεφαλαίο. Αφορά τη ολογική σκέψη. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ça vote tout seul. C'est bien, on a une machine qui vote toute seule. Μια, un μηχάνημα fait να ψηφίζει από μόνο του. 27 ψηφίσαντες, 23 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Έλλης. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Περνάμε στην έκθεση Κοτινή. Οργάνωση ε, της... Ε, έρευνας για, το εργατικό δυναμικό στην κοινότητα, δειγματοληπτική έρευνα. Ζαν Λουί Κοτίνη. Κοινότητα, υπάρχει ακόμη η ευρωπαϊκή κοινότητα. Τέλος πάντων, ποια κοινότητα, δεν ξέρουμε για ποια κοινότητα πρόκειται. Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 2 και 3. Ο εισηγητής είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τρεις αποχές, χωρίς αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικέ σκέψει, τροπολογία 1 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Τρεις κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. «28 ψήφισαν, 28 είμαστε, 27 ψήφισαν όμως» περίεργο. Μήπως θα μπορούσαμε να ξυπνήσουμε τον 28 τον 28ο ή δεν θέλει να ψηφίσει. Τέλος πάντων, λίγη ψηφοφορία, ψήφισαν 24 υπέρ και 3 κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια στο Ζωάν Λουί Κοτινή. Έκθεση Utah Hawk. Α, είπαμε να την αναβάλουμε αυτή την ψηφοφορία. Όχι μόνο για την έμψα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ασφάλεια της Ναυσιπλοεία. Αυτό αναβάλουμε, το 27 δηλαδή, το 23 συγγνώμη, αλλά ψηφίζουμε για το 24, τη Europol. Τον Οργανισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωση για τη συνεργασία σχετικά με την επιβολή του νόμου και την κατάρτιση. Α, περίπλοκα τα πράγματα, για τη αστυνομία μιλάμε. Τροπολογία 5 και τροπολογία 11. Θα τις ψηφίσουμε μαζί. Ναι μεν, αλλά σε τρία τμήματα. Πρώτα το κοινό τμήμα των δύο τροπολογιών 5 και 11. Η συγκέντρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τρεις κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο, ψηφίζουμε την προσθήκη στον προϋπολογισμό του οργανισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη δεύτερη ψηφοφορία. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμη αυτός που κοιμάται 28ος. 12 υπέρ 14 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε και στην τρίτη ψηφοφορία. Ισχύει. Προφορική τροπολογία της συγγήτριας για διαγραφή του and accounting. Ποιος είναι υπέρ της διαγραφής. Κατά. 2. Αποχές. Εγκρίνεται με μία αποχή. Αυτά για τις δύο τροπολογίες. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 6 της συγκεκριτρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μία ψήφο κατά. Για την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Έχουμε τρει τροπολογίες Θα Μπορούμε να τι ψηφίσουμε μαζί. Α, συγγνώμη, έχω ξεχάσει την αιτιολογική σκέψη. Τροπολογία 4, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με τρει ψήφου κατά. Τώρα για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματο. Να ψηφίσουμε μαζί τι τροπολογίε 1, 2 και 3 τη συγκεντρία. Ναι, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Μία ψήφο κατά εγκρίνεται. Ε, μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί όλες τις τροπολογίες της κυρίας Χολμάιερ. Η συγκέντρη είναι υπέρ. Έχουμε και προφορικές ενδιάμεσα, αλλά φαντάζομαι ξέρουμε όλοι γιατί μιλάμε. 7, 8, 9 και 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με τρεις ψήφους κατά και μία αποχή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Σαλβαντόρ δίνει σφυριά στο μηχάνημα, αλλά ο κοιμισμένος εξακολουθεί να κοιμάται. Από τους 28 λοιπόν ψήφισαν μόνο 27, 23 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας την κυρία Γιούτα Χάουκ. Έχουμε μεταφορές πιστώσεων. Μπορεί κάποιος να αντικαταστήσει τον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Λαβία, για τις μεταφορές. And, ε, Λαβία. Okay. Donc, Κοιτάξτε, όλα μας τα εξήγησαν σήμερα το πρωί από ό,τι φαίνεται. Τι ωραία, όταν δεν προεδρεύω εγώ όλα πάνε καλά. Λοιπόν, αρκεί να ψηφίσουμε τότε. Θα ψηφίσουμε το ένα μετά το άλλο λοιπόν. Είναι πιο απλό έτσι. Το 10, 16, ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Μία αποχή. Δεκτό. Δεκ 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ένας κατά δύο κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεκαοκτώ, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Αποχές. Δεκτό. 19. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δύο κατά, αποχές δεκτό. Το 21, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, μία αποχή. Για τα υπόλοιπα τμήματα μας άφησε μια κληρονομία ο κ. Λαβία από το πρωί. Τα εξήγησε όλα. Και είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Λοιπόν για τα κτίρια δεν το συζητάμε οπότε δεν ψηφίζουμε πλέον. Δεν έχουμε καμία άλλη ψηφοφορία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τελειώσαμε. Όχι. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε αρκετά σημεία να εξετάσουμε ακόμα, ελπίζω σύντομα. Το 8 για τους ιδίους πόρους και το MFF. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε αρκετά στους συντονιστές και χθε στην ομάδα επαφής. Έχουμε ένα εισηγητή εδώ μαζί μας, τον Ζων Λουκ. Να παρουσιάσω την κατάσταση ως εξής και θα με ελέγξει. Προχωρήσαμε λοιπόν στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η οποία με μεγάλη πλειοψηφία, πέραν της απόλυτης, επιβεβαίωσε τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου που εκφράστηκε από μένα και τον κύριο Σούλτς την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή αυτήν την μήνυ συνάντηση κορυφής σύμφωνα με το άρθρο της συνθήκης για τις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις. Στα πλαίσια αυτού του ψηφίσματος τώρα στείλαμε ορισμένα πολιτικά μηνύματα και διευκρινίσαμε ότι η τελική ψήφος, η οποία είναι η μοναδική που έχει μία νομική σημασία και που θα αφορά τη συνολική συμφωνία και θα καλύψει και τον κανονισμό MFF, και την διαθεσμική, ε, διοργανική μάλλον συμφωνία. Αυτό θα γίνει αργότερα, μετά τις διακοπές και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πότε ακριβώς. Αλλά αυτό θα γίνει τη στιγμή κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι βέβαιο ότι ε, το δεύτερο τμήμα του διορθωτικού για τις πληρωμές του 2013, 3 εκατομμύρια, θεωρείται δεδομένο. Και από την άλλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι επίσης βέβαιο ότι θα διεξαφούν σωστά οι διαπραγματεύσεις για τα νομοθετικά κείμενα. ο εκπρόσωπος της Λιθουανικής Προεδρίας, ο οποίος ήταν παρόν στην διάσκεψη των Προέδρων την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι υπάρχουν γύρω στις 70 προτάσεις κανονισμού που θα πρέπει να υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας επί τη βάση των νομικών βάσεων των πολιτικών που άπτονται του προϋπολογισμού. Εξάλλου, στην συνάντηση των συντονιστών διαπιστώσαμε ότι όλοι οι συντονιστές συμφωνούν έτσι ώστε για το τέλος της διαδικασίας, την υιοθέτηση δηλαδή του MFF και μετά την υιοθέτησή του εφόσον γίνει εν αυτό υποθέτουμε επί τη βάση της ψηφοφορίας που έγινε στην Ολομέλεια. Είναι επιθυμητό το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών σε συνεργασία με την Επιτροπή ΑΦΚΟ να καταλήξουν στα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα, μαθήματα αν θέλετε, ε, μετά το τέλος αυτής της διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση αυτή ήταν απογοητευτική. Ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρενέβη στον καθορισμό του δημοσιονομικού πλαισίου των επομένων 7 ετών είναι ιδιαιτέρως απογοητευτικό, προκαλεί δυσθυμία και είναι ασύμβατο κατ' εμέ τουλάχιστον με το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Το γράμμα έγινε τύπη σεβαστό, αλλά όχι το πνεύμα. Από ό,τι φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ε, εξελίχθηκαν τα πράγματα ε, οδηγεί στο να μειωθεί σημαντικά η δημοσιονομική εξουσία του Κοινοβουλίου και σε επίπεδο ετησίου ε, δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί εφόσον τα περιθώρια είναι πάρα πολύ χαμηλά ε, στην ουσία είναι σαν να έχουμε προαποφασίσει ε, το ύψος των επομένων προϋπολογισμών, ως εκ τούτου το περιθώριο διαπραγμάτευσής τους είναι ελάχιστο. Και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι διαπραγματεύσεις απομείωσαν την εξουσία, την αρμοδιότητα, τη συνομοθετική του Κοινοβουλίου και των υπολείπων επιτροπών. Όπως είπαμε υπάρχουν 70 διαπραγματεύσεις οι οποίες τρέχουν, αλλά ε, ξέρουμε ότι σε κάποια βασικά θέματα που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες επίπεδο κόστους ε, πολιτικές, μεταφορές, γεωργία βέβαια, Ευρώπη 2020, Εράσμους για όλους, Ξέρουμε λοιπόν ότι για όλες αυτές τις πολιτικές η Ιρλανδική Προεδρία και τώρα η Λιθουανική Προεδρία η οποία διαπραγματεύεται με τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου εκφράζουν την άποψη ότι ό,τι έχουν πει μέχρι τώρα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8 η Φεβρουαρίου δεν αλλάζουν με τίποτα, είναι χαραγμένα στην πέτρα και ως εκ τούτου από εδώ και πέρα η νομοθετική εξουσία ουσιαστικά μεταφέρθηκε στο Συμβούλιο. Ένα όργανο ε, του οποίου βέβαια την ύπαρξη αναγνωρίζει η Λισαβόνα αλλά και στο οποίο η συνθήκη της Λισαβόνας απαγορεύει να έχει νομοθετικό ρόλο. Πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό και, ε, και θεσμικό ακόμα πρόβλημα. Βρεθήκαμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση πλέον που το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του εδώ και λίγες μέρες απεδέχθη το αποτέλεσμα για το δημοσιονομικό πλαίσιο τουλάχιστον. Θα δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο νομοθετικό. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζουμε ότι το σύνολο των συμμετεχόντων αναγνώρισαν ότι δεν μπορούμε εμείς να μην καταλήξουμε στα αποτελέσματα και στα συμπεράσματα αυτής της κατάστασης και ότι είμαστε ηθικά, δεοντολογικά υποχρεωμένοι αλλά και πολιτικά υποχρεωμένοι να το ε, εκφράσουμε επίσημα και να ε, ε, δώσουμε συστάσεις αν θέλετε επίσημες προς το επόμενο κοινοβούλιο στο επερχόμενο κοινοβούλιο έτσι ώστε ε, ο ρόλος του να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της αναθεώρησης η οποία προβλέπεται στη Συμφωνία MFF από το 16 και το 17. Αυτό θα γίνει με τον εξής τρόπο, με την εξής μορφή. Πρώτον, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε την έκθεση της ΑΦΚΟ, η ΑΦΚΟ είναι υπεύθυνη, ε, για την διοργανική συμφωνία. Αυτή η διοργανική συμφωνία είναι κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα η ΑΦΚΟ. Ε, ταυτόχρονα θα δώσουμε εμείς μια γνωμοδότηση προς την ΑΦΚΟ και θα προτείνουμε και τροπολογίες εφόσον το επιθυμούμε γνωρίζοντας όπως όπως και να έχουν τα πράγματα η έκθεση ΑΦΚΟ είναι πάρα πολύ συνοπτική ένα άρθρο είναι, λέει ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει την διοργανική συμφωνία, αλλά μπορούμε εμείς στις αιτιολογικές σκέψεις να προχωρήσουμε σε τροπολογήσεις. Οι εισηγητές για το MFF είναι οι υπεύθυνοι που θα μας προτείνουν ε, πιθανές τροπολογίες. Δεύτερον, με τους συντονιστές αποφασίσαμε να συντάξουμε μία έκθεση πρωτοβουλίας ε, για την οποία θα επιφορτιστεί ο εισηγητής και σε συνεργασία με την ΑΦΚΟ θα δούμε τώρα πώς θα το μοιράσουμε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 50 και τα λοιπά, θα τα διευκρινίσουμε. Όμως, στόχος μας είναι αμέσως μετά την τελική ψήφο μετά την τελική ψήφο για να μην υπάρξει σύγχυση αν θέλετε για την ψηφοφορία οι συγητές θα συντάξουν μια έκθεση πρωτοβουλίας για τα συμπεράσματα, τα μαθήματα από την ακολουθούμενη διαδικασία και για τις πιθανές βελτιώσεις τις οποίες πρέπει να ζητήσει, να απαιτήσει και να πετύχει ήδη στα πλαίσια της επόμενης αναθεώρησης έτσι ώστε η έκθεση αυτή να ολοκληρωθεί και να υιοθετηθεί από την Ολομέλεια πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Ε, στις αρχές του 2014 γιατί θα μπορούσε κανείς να φοβηθεί ότι λόγω ακριβώς των επερχομένων εκλογών από την άνοιξη, τις αρχές της άνοιξης και μετά θα ασχολείται ο κόσμος με άλλα πράγματα και όχι να κάθεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο συμφωνήσαμε με τους συντονιστές. Αυτά. Δεν ξέρω, έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, μια κάποια συμπλήρωση σε αυτό το πλαίσιο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Καλώς, σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο. Σημείο 17. Έκθεση Κατρίν Τροτμάν που μας κάνει την τιμή και μας δίνει τη χαρά της παρουσίας της. Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα είμαι πολύ λακωνική γιατί γνωρίζετε το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής. Μοιάζει με την προηγούμενη και μάλιστα κάποια σημεία έχουν ήδη ξεπεραστεί γιατί τότε προσπαθούσαμε να συμβάλλουμε στην στρατηγική της Επιτροπής μας για κατάλληλο προϋπολογισμό, ικανοποιητικά κονδύλια. Όλα αυτά τα θέματα πια είναι παροχημένα μετά τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό και θα αναγκαστώ να καταθέσω κάποιες διορθωτικές τροπολογίες. Επί της ουσίας θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο γιατί ξέρω ότι υπάρχει συνένεση στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η οικονομική του συμμετοχή στον προπολογισμό της Ένωσης και στην προσπάθεια να εδραιωθούν οι προσπάθειές τους και να εξηγιαθούν τα οικονομικά τους, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κάτι που δεν ε, έχει ακόμη συζητηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Επί της ουσίας πάντως δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια. Παρά μόνο για το σημείο 7. Για τους ιδίους πόρους. Ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, ιδιαίτερα μετά τόσα ακούσαμε για τις, για συνέπειες του front-loading και του back-loading στις δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτά εν ολίγης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όσα έχω ήδη πει για την προηγούμενη έκθεση. Πολύ ωραία. Χθες Είμαι προσκεκλημένος στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση για να λάβω μέρος σε μια συνεδρίαση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Βουλής με το γραφείο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Λιθουανικής Βουλής. Οι Λιθουανοί είπαν ότι συμφώνησαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρώτη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση του άρθρου 13, δηλαδή για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Οπότε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και αυτή την υπόθεση. Αρμόδια βέβαια καθήλ είναι κυρίως η Επιτροπή ΕΚΟΝ, αλλά και εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα. Η Κατρίν Τροτμάν. Κάτι που δεν λέω στην έκθεση, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω εδώ. Είχαμε πολλές κοινέ ε, συνεδριάσεις με την ΕΚΟΝ και χαίρομαι γι' αυτό. Καλό θα ήταν όμως πριν τη διακοινοβουλευτική αυτή συνεδρίαση να συντονιστούμε λίγο με την ΕΚΟΝ και να έχουμε διαβουλεύσεις έγκαιρες με την ΕΚΟΝ ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στη διαμόρφωση της ε, θέσης. Ακριβώς επειδή έχουμε πολύ συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο. Και αυτό θα πρέπει να το διατρανώσουμε. Ιδιαίτερα τη στιγμή που οι εθνικές βουλές από ό,τι φαίνεται μπαίνουν στον πειρασμό να αναλάβουν αυτές την κατάσταση στα χέρια τους, στα ενία της κατάστασης. Είναι χρήσιμο λοιπόν να συντονιστούμε με την ΕΚΟΝ. Και καλό θα ήταν να, να το επισημάνουμε, γιατί νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολόκληρο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι για την έκθεση της Κατρίν Τροτμάν η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει στις 30 Αυγούστου. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Οικονομική Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενώ στην Ολομέλεια το θέμα θα περάσει στη δεύτερη Ολομέλεια το Οκτωβρίου και όπως μας είπε σωστά η Κατρίνη Τωροτμά θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς μαζί με την ΕΚΟΝ για να συντονίσουμε τη θέση μας ό,τι αφορά την προετοιμασία της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης του άρθρου 13. Άλλωστε θα είμαστε στη των ταυτόχρονα με την ΕΚΟΝ. Ε, είμαστε μάλλον ταυτόχρονα με την ΕΚΟΝ, αλλά τότε ε, είχαμε ζητήσει να συναντηθούμε και με τα μέλη τη ΕΚΟΝ, αλλά το επιχείρημα των μελών τη ΕΚΟΝ ήταν ότι η αντιπροσωπεία του πήγε στη Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με του ομολόγου των ΗΠΑ, όχι για να ξαναδεί εμά. Αυτά. Αν δεν υπάρχουν άλλε παρατηρήσει, να περάσουμε σε ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλέ στον Σαλβαντόρ, Γκαρίγκα, το σημείο 15 δηλαδή. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για τη Λομβαρδία στην Ιταλία. Ο Σαλβαντόρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ λακωνικός. Η επιχειρηματολογία είναι η ίδια. Το θέμα αφορά κάποιες ε, δράσεις στη Λομβαρδία για τις ευφυείς τηλεπικοινωνίε. Και οφείλεται στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Είχαμε εξαιτία τη παγκοσμιοποίηση και τη κρίση 529 απολύσει στι εταιρείε τηλεπικοινωνιών στη Λομβαρδία. Τελικά 480 έμειναν χωρίς ε, δουλειά. Γι' αυτό και χρειάστηκαν κάποια μέτρα και κονδύλια από το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Η Λομβαρδία είναι από τι πιο ευημερού περιοχέ και πιο βιομηχανισμένε περιοχές της Ιταλίας με ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογία. Οι σχετικές όμως προηγμένες τεχνολογικές εταιρείε επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Γι' αυτό και προτείνεται η κινητοποίηση αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής για τη Λοβαρδία. Προσπαθώντας να αντισταθμίσουμε την ε, θέση του Συμβουλίου να μπλοκάρει τη ρήτρα οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς ελάχιστη ευαισθησία έχει δείξει το Συμβούλιο, όπως δείχνει η απόφαση της 8 Φεβρουαρίου, για να, μειωθεί, ε, να μειωθούν δραστικά η πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων για τη νέα περίοδο χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ενώ περιπτώσει σαν αυτή τη Λομβαρδία δείχνει πόσο σημαντικό είναι το ταμείο αυτό και πόσο συγκεκριμένη είναι η βοήθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους είτε λόγω της οικονομικής κρίσης είτε λόγω της παγκοσμιοποίησης. δεν έχει ιδιαιτερότητα στο θέμα αυτό. Είναι χαρακτηριστικό, χαρακτηριστική περίπτωση για την οποία ζητούμε συνήθως κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Και εγώ είμαι υπέρ. Ένα σύντομο σχόλιο, λέει η ΕΙΔΕΡ. Στο τελευταίο τριμερή διάλογο φτάσαμε ευτυχώ ε, στη συμφωνία ώστε να ληφθεί υπόψη και το κριτήριο της οικονομικής κρίσης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εξού και οι τροπολογίες, οι διορθωτικές που θα καταθέσουμε. Φυσικά και είμαστε και εμεί υπέρ της κινητοποίηση του Ταμείου. Λέμπρα. Χρονοδιάγραμμα. 29, Ιουλίου, ε, 29 συγγνώμη, Αυγούστου λίγη προθεσμία για τις τραπολογίες, 18 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Απασχόλησης και εμείς το ίδιο ενώ το θέμα θα πάει στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου ή την πρώτη ή τη δεύτερη, δεν είναι σίγουρο ακόμη. Σημείο 14. Ο Νταμινίκ Κρικέ θα μας μιλήσει για την κινητοποίηση του ίδιου ταμείου, αλλά για άλλο θέμα, την αυτοκινητοβιομηχανία το Μάζο Ετομόβιλε της Ιταλίας. Περνάμε στο Πεδεμόντιο και στην Τοσκάνη σε ένα αντίστοιχο θέμα. Δεν θα επανέλθω στις παρατηρήσεις και τα παράπονα του Σαλβαντόρ, τα οποία συμφωνώ. Μιλάμε για αυτοκίνητα, έχουμε μια κρίση μέσα στην κρίση. Δηλαδή, στο γενικότερο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης γνωρίζουμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία που αντιμετωπίζεται και με άλλους τρόπους βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εταιρεία Ντετομάζο είναι γνωστή σε αυτούς που αγαπούν τα αυτοκίνητα γιατί για πάρα πολλά χρόνια ε, παρήγαγε ένα ιδιαίτερα ακριβό και πολυτελές αυτοκίνητο, προσπάθησε να προσαρμοστεί, απορρόφησε ένα τμήμα της ε, επιχείρησης Πινιμφαρίνα, πέρασε από 250 σε 1000 τόσους ε, εργαζομένους και αυτό στάθηκε μοιραίο η προσπάθεια για αυτοκίνητα ευθυνότερα δεν ακολουθήθηκαν από θετικά αποτελέσματα, απορροφήθηκε από την κρίση, αυτές οι προσπάθειες έγιναν το 8, 9 και 10, πήγαν χάλια τα πράγματα και τώρα οδηγηθήκαμε σε πτώχευση που ε, ανακοινώθηκε τον Απρίλιο και στο τέλος του 12 δικαστικά κατακυρώθηκε. Η επιχείρηση όπως είπα δημιουργήθηκε η τελευταία μετά από την συνεργασία ανάμεσα στην επιχείρηση Ντετομάζο και στην επιχείρηση Πινιμφαρίνα αφορά 1030 εργαζομένους. Σύμφωνα με την νομοθεσία και όπως γνωρίζουμε οι Ιταλικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν εν πάση περιπτώσει μια πρωτοβουλία η οποία είναι αποδεκτή, θεμητή και ζητείται από την Επιτροπή μας να εγκρίνουμε την παρέμβαση του Ταμείου αυτού έτσι ώστε να λάβει υπόψη το 50% της παρέμβασης, δηλαδή 2.584 και κάτι ψηλά, χίλια εκατομμύρια ευρώ, χιλιάδες ευρώ μάλλον. 2 εκατομμύρια 500 περίπου χιλιάδες ευρώ. Ευχαριστώ κύριε Ερικέ πράγματι για την δική μας γενιά ε, είχε τρομερό γόετρο η επιχείρηση δεν το μάζω, και ένας γιος της οικογένειας είχε σκοτωθεί σε, στο ράλι του Μοντε Κάρλο χτυπώντας ένα αυτοκίνητο, οδηγώντας ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχουμε ένα πρότυπο εδώ υπόδειγμα της εφαρμογής των δυνατοτήτων του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του οποίου αναγνωρίζουμε τώρα πλέον το ενδιαφέρον, το οποίο διέφυγε βέβαια του Συμβουλίου δεν διέφυγε ημών βέβαια. Λοιπόν, η προθεσμία είναι η 29η για τις τροπολογίες Αυγούστου και όπως και για την προηγούμενη περίπτωση οι ψηφοφορίες θα γίνουν στην Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 18 Σεπτεμβρίου με πιθανή ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον μήνα Οκτώβριο. Περνάμε τώρα λοιπόν στο 18. Έιντα. Ε, χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη-μέλη με ιδιαίτερες δυσκολίες χρηματοοικονομικές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω το στόχο αυτής της ε, γνωμοδότησης με λίγα λόγια. Πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών αλλά αφορά τη φιλοσοφία ουσιαστικά των ε, Ταμείων Συνοχής. Λέμε γιατί υπάρχουν τα Ταμεία Συνοχής και γιατί θεσπίστηκε η πολιτική συνοχής. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι τα Ταμεία Συνοχής ε, δημιουργήθηκαν ως έκφραση αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως των πιο ευημερουσών περιοχών προς τις λιγότερο ε, ευημερούσες, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια εποχή κρίση αυτή που βιώνουμε τώρα και μια εποχή που πολλές περιφέρειες δεν έχουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς κονδύλια για να επενδύσουν στις πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, είναι αναμενόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσουν τροποποιώντας τις διατάξεις ε, και λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση. Δύο είναι οι λύσεις που προτείνω εγώ στην νομοδότηση. Δύο τρόπους δράσης μάλλον. Καταρχήν το είναι συν τρία που είναι ο κανόνας που έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει το ενίσυν 3 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μια και αυτή θα είναι η γραμμή για το μέλλον να εφαρμοστεί ο κανόνας ενίσυν 3 και για το 2013 που ούτως ή άλλως έγινε για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι οι μόνες χώρες που έχουν προβλήματα χρήσης των ε, κονδυλίων της συνοχής. Ούτε είναι οι μόνες χώρες που ε, αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρέ δυσκολίε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα και του κανόνε αποδέσμευση. Γι' αυτό θα έλεγα όλα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τον κανόνα νησιν 3 και πριν την επόμενη προγραμματική περίοδο, ήδη δηλαδή από το 2013. Δεύτερη γραμμή που προτείνω είναι ότι αν θυμάστε ε, ήδη τροποποιήθηκε κάποια κράτη-μέλη το ποσοστό συγχρηματοδότηση. γιατί εξαιτία τη κρίση πολλέ περιφέρειε δεν μπορούν να πληρώσουν το μερίδιο της χρηματοδότηση που τους αντιστοιχεί. Και κάποιες χώρες που επειδή βρισκόταν υπό ευρωπαϊκή εποπτεία και ακολουθούσαν προγράμματα διάσωσης και μνημό, εφάρμοζαν μνημόνια, για τις χώρες αυτές προβλέφθηκε μια αλλαγή του ποσοστού χρηματοδότησης για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα τα ταμεία της συνοχής. Πιστεύω ότι αυτό το μέτρο θα πρέπει επίσης να διευρυνθεί, να επεκταθεί και σε άλλες χώρες, γιατί και εδώ δεν είναι δυστυχώς μόνο αυτές οι χώρες που έχουν προβλήματα με τα κονδύλια της συνοχής και την ε, αδυναμία τους να καλύψουν το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Γιατί και οι χώρες που έχουν υπερβολικό έλλειμμα που είναι το κριτήριο που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο και γνωρίζουμε ποιες είναι οι χώρες, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Αυτά τα δύο μέτρα λοιπόν προτείνω στην γνωμοδότησή μου και περιμένω τα σχόλιά σας και ελπίζω φυσικά όταν έρθει η στιγμή της ψηφοφορίας να υπερψηφίσουμε την γνωμοδότηση γιατί πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τα κράτη-μέλη. Yeah. Ε, Ευχαριστώ, Αιντέρ. Έχετε μήπως παρατηρήσεις, συστάσεις προς την εισηγήτρια. Όχι. Οπότε να υπενθυμίσω ότι για την γνωμοδότηση της Αιντέρ η προθεσμία και εδώ για την κατάθεση τροπολογιών λήγει 29 Αυγούστου στις 6. Θα ψηφίσουμε στις 18 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για να επιδώσουμε την πρότασή μας στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα ψηφίσει στις 23 Σεπτεμβρίου ώστε να περάσει το θέμα στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ένα και μόνο σημείο μας απέμεινε, το σημείο 16 Η γνωμοδότηση που θα πρέπει να επιδώσουμε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάκτης γνωμοδότησης ήταν ο Αλεξάνδρ Άλβαρο που είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο. Χαίρομαι γιατί τα νέα για την κατάσταση υγείας του είναι πολύ θετικά και αισιόδοξα, αλλά φυσικά δεν έχει αναρρώσει ακόμη για να είναι μαζί μας. Αν δεν κάνω λάθος, θα έρθει να πάσει στιγμή ο κύριος Μιούλτερ. Αλλά πώς, με τα πόδια, με ποδήλατο, με κανένα αυτοκίνητο το μάζω Εν πάση περιπτώσει, όσο τον περιμένουμε, να σας πω ποια θα είναι η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών. Η γνωμοδότηση αναλύει το κατά πόσο η η ύπαρξη πολλών εδρών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβαρύνει τον προπολογισμό και αν συμφέρει περισσότερο η ενιαία έδρα. Τεράστιο το suspense αυτή τη γνωμοδότηση όσο περιμένουμε τον κύριο Μούλτερ. Η κατάθεση των τροπολογιών θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι το 16 Ιουλίου. Πολύ σύντομη προθεσμία λοιπόν. Οπότε αν θέλετε να προτείνετε πολλές νέες έδρες, έχετε μέχρι 16 Ιούλιο να το κάνετε. Θα ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή, στις 17 να ψηφίσει η αρμόδια καθήλια Επιτροπή. Ο Γκέρον. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Γιάννη Μιούλτερ, αλλά όσον τον περιμένουμε, να πω δύο λόγια και εγώ. Καταρχά, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο Αλεξάνδρου Άλβαρο ήταν σε θέση να καταρτήσει την έκθεση αυτή. Αυτό ελπίζω να σημαίνει ότι θα τον δούμε σύντομα και προσώπους εδώ στην Επιτροπή. Και χαίρομαι επίση ε, γιατί η έκθεση φαίνεται να κινείται προ σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σύντομη. Και όλε αυτέ οι πραγματοποιήσει ασφαλώ είναι πάρα πολύ σύντομε στην έκταση. Δεν ξέρω κατά πόσον συνάδελφοι σκοπεύουν να καταθέσουν τροπολογίε για να τονίσουν πιο πολύ βασικά τα αμυγό χρηματοοικονομικά θέματα, τα θέματα προπολογισμού της γνωμοδότησης. Να ξεκαθαρίσουμε στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου ότι έχουμε σωστά και αξιόπιστα αριθματικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό για τις δύο έντρες. Αυτά λοιπόν σκοπεύουμε να καταθέσουμε ως τροπολογίες. Ελπίζω να μας βρείτε, να συμφωνήσετε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή Προπολογισμών έχει ως ρόλο να διευκρινίσει τα στοιχεία αυτά και να κάνει τους ακριβέστερους δυνατούς υπολογισμούς. Πόσο στοιχίζει το ισχύον σύστημα και σε περίπτωση που επιλεγεί ενιαία έδρα, ποιο θα είναι το κόστος της μίας και μόνο έδρας. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν κάποιες οικονομίες. Από αυτή την άποψη, οι εκτιμήσεις που ακούσαμε δίστανται πολύ σημαντικά. Έφτασε η βεντέτα μας, ο Γιάνν Μίλντερ. Θα του δώσω λίγο χρόνο για να καθίσει και θα του ζητήσω να μας κάνει μια ενημέρωση για την γνωμοδότηση που ανέλαβε από τον κύριο Άλβαρο και που αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες τη, το διπλής έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αν επί τη ευκαιρία έχει κάποιες ειδήσει για τον Άλβαρο, μα ενδιαφέρει πολύ. Να σας πω ότι τον περιμένουμε το Σεπτέμβριο ήδη. Very good. On the... Ωραία. Για το πρόβλημα το οποίο αναφέρατε σε ό,τι αφορά την έντρα του Κοινοβουλίου. Είμαι Ολλανδός. Και ένα πράγμα στην πολιτική της Ολλανδίας ενώνει όλα τα κόμματα. Και αυτό είναι το εξής. μία και μόνη έδρα για το Κοινοβουλίο. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψη που εκφράζει ο Αλεξάνδρα Άλβαρο. Και αυτό αποτελεί αν θέλετε και το ζουμί της έκθεσης. Θα παρουσιάσουμε και κάποιες επιπρόσθετες τροπολογίες για την έκθεση. Θα διευκρινίσουμε με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια στοιχεία, αλλά νομίζω ότι η γενική σύσταση είναι ότι είναι προτιμότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία και μόνο έδρα. Και έχει περάσει και η ώρα, ξέρετε, και δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρος από αυτό. Μάλιστα. Ο ρόλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών είναι εδώ να διευκρινίσει τα αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχει μια πολιτική θέληση. Η πολιτική θέση θα εκφραστεί από την Συνταγματική Επιτροπή. Εμείς έχουμε το αριθμητικό στοιχείο. Γιατί διαβάσαμε αριστερά και δεξιά πολύ διαφορετικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς. Και μερικές φορές είναι και άλλο πρόσελα τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών αφορά μόνο τα αριθμητικά στοιχεία. Αυτό είναι ο ρόλος μας για ένα πολύ λεπτό θέμα, το οποίο γνωρίζουμε, αλλά η πολιτική συζήτηση δεν θα γίνει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, αλλά στην Συνταγματική Επιτροπή, η ΑΕΔΕΡ. Ένα από τα σχόλια τα οποία θα ήθελα να κάνω ήταν ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή γιατί είναι προφανές υπάρχουν διαφορετικές μελέτες που μας δίνουν ε, κάποιους αριθμούς αλλά και τους αντίθετους τους είναι εντελώς υποκειμενικοί. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα λοιπόν είναι ένα θέμα προσωπικό για κάθε ένα βουλευτή και γι' αυτό νομίζω ότι σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να είμαστε επακριβέστατοι σε σχέση με τους αριθμούς, να δώσουμε τους πιο αντικειμενικούς αριθμούς και ο καθένας να αποφασίσει αν δημοσιονομικά μπορεί να είναι υπέρ ή κατά της ενιαίας έδρας. Να θέσω ένα ερώτημα. Μιλάμε για την μοναδική έδρα ο τίτλος αναφέρεται στα ευρωπαϊκά όργανα. Γνωρίζουμε ότι μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τι γίνεται με το Λουξεμβούργο. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε στο Στρασβούργο ενώ ε, η δουλειά μας γίνεται στις Βρυξέλλες. Αλλά όμως υπάρχει και στο Λουξεμβούργο και αν η απόφαση για μια ενιαία έδρα λαμβάνει υπόψη το Λουξεμβούργο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας γιατί το να μεταφέρουμε το Λουξεμβούργο εδώ που έχει όλα τα γραφεία είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει ένα κόστος και πρέπει να ληφθεί υπόψη στον καθορισμό του κόστους της ενιαίας έδρας. Και ένα τελευταίο σχόλιο ότι ανεξαρτήτως της τελικής θέσης και το εάν το κοινοβούλιο αυτό επαναλάβει για μια ακόμη φορά ότι θέλουμε να συγκεντρώσουμε τις εργασίες μας στις Βρυξέλλες και ας υποθέσουμε ότι το Συμβούλιο δέχεται και να γίνει αυτή η κίνηση. Τότε θα πρέπει να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ήταν και πηγαίνει στο Στρασβούργο ακριβώς λόγω του συμβόλου που αποτελεί αυτή η πόλη ε, και σύμβολο συμφιλίωσης και δεν μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση χωρίς τη συμφωνία των γαλλικών αρχών και προσπαθώντας να βρούμε και μια διαφορετική χρήση για το κτίρια τα οποία είναι εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό. Λοιπόν, αν τελικά πάρουμε την απόφαση ότι πρέπει να δουλεύουμε μόνο στις Βρυξέλλες, όλα αυτά θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί σωστά και να υπάρξουν σωστές και χρήσιμες ιδέες για το τι θα γίνει με τα κτίρια του Στρασβούργου. Δεν μπορούμε να κλειδώσουμε και να σκοθούμε να φύγουμε. Η Κατρίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μπω στη συζήτηση επί της ουσίας. Θα ήθελα και εγώ όπως οι συνάδελφοι, άλλωστε έχω μαζί με τη Σιλβίγκη Γιώμ καταθέσει μια τροπολογία σχετικά με την ανάγκη να έχουμε πραγματικά αντικειμενικούς αριθμούς. Σχετικά λοιπόν με τους αριθμούς να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι αριθμοί αυτοί θα πρέπει να είναι ακριβείς, όπως είπα. Γιατί οι εμπειρίες που έχω γύρω από τη συζήτηση αυτή εδώ και αρκετά χρόνια είναι ότι μπορεί κανείς να κάνει υπολογισμούς με διαφορετικούς τρόπους. Χρειάζονται λοιπόν επακριβείς αριθμοί για τον υπολογισμό της λειτουργίας των κτηρίων μας. Να περιλάβουμε και το κόστος της απόκτησης, το οποίο μπορεί να επιβαρύνει ακόμα και για μία μακρά χρονική περίοδο ε, το ε, προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και που επηρεάζει ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό αυτό και μιας και μιλάμε για τις δημοσιονομικές προοπτικές σε σχέση με τα κτίρια πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο γιατί έτσι υπολογίζουμε το κόστος λειτουργίας ε, ενός κτηρίου, το κόστος απόσβεσης ε, αυτό θα είναι πιο συγκεκριμένο από κάποιες θεωρητικές αναλύσεις σε σχέση με πιθανές μελλοντικές προβολές για, την οικολογική, για τον οικολογικό ισολογισμό αν θέλετε του κτηρίου. Και ταυτόχρονα η Επιτροπή μας θα πρέπει να προσπαθήσει να δει ποιε είναι οι προβλέψεις ε, για τα κτίρια αυτά και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη χρήση του στο μέλλον και αναφέρομαι εδώ σε κόστη όπως το κόστος συντήρησης, γιατί αν θέλουμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται σε σχέση με το κόστος των κτηρίων. Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να προσθέσω σε αυτή τη συζήτηση, έτσι ώστε η συζήτηση όταν γίνει να γίνει γνωρίζοντας ε, ε, ε, ακριβώς τα πράγματα. Μία μικρή παρατήρηση. Η συνθήκη λέγει ότι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το Στρασβούργο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις έδρες εργασίας. Παρακαλώ μην το ξεχνάτε, πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια αυτό που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 11, ε, ε, του 91 συγγνώμη, ε, δεν υπήρχε η έννοια της έδρας, υπήρχε μόνο αναφορά στους χώρους εργασίας, στους τόπους εργασίας και ένα από τα προβλήματα της έκθεσης αυτό είναι ότι σήμερα μία έδρα υπάρχει το Στρασβούργο. Λοιπόν, δεν αναφέρομαι στα υπόλοιπα, αναφέρθηκα απλά σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι στον τίτλο της έκθεσης ε, του ΑΦΚΟ λέγεται στα αγγλικά ο καθορισμός της ένδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε αναφερόμαστε σε πολλές έδρες. Όταν όμως μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό καθεαυτό, νομικά έχει μία έδρα με πολλούς τόπους εργασίας. Αυτό που είπε η Κατρίνη είναι αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι να ξεκαθαρίσουμε τους αριθμούς και όπως το είπε και η Ιντερ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ε, το Λουξεμβούργο, το τι κοστίζει το Λουξεμβούργο σε επίπεδο οικονομικό και διοικητικό. Δεν έχουμε Λουξεμβουργιανούς ανάμεσά μας, αλλά ίσως για να ζωηρέψει η συζήτηση να προσκαλέσουμε στην επόμενη συζήτηση την κυρία Λούλινγκ η οποία θα εμπλουτίσει ιδιαιτέρως και την ουσία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα όπως και σε πολλά άλλα. Λοιπόν, θυμίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική, δύσκολη, ευαίσθητη και ρόλος μας σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι να δώσουμε αντικειμενικά στοιχεία αριθμητικά έτσι ώστε αργότερα οι πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν να λαμβάνονται γνωρίζοντας πραγματικά την κατάσταση. Συγγνώμη, Γιάννα. Ευχαριστώ. σπάνιο, αλλά συμφωνώ σχεδόν με όλες τις παρατηρήσεις. Να λάβουμε υπόψη και το κόστος του Λουξεμβούργου. αλλά δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο με το Στρασβουργό, δεν έχουμε το ίδιο τσίρκο της μιας εβδομάδας το μήνα, όπως γίνεται με το Στρασβούργο, είναι σχεδόν διοικητική η έδρα. Και συμφωνώ, θα πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος, γιατί αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Όπως είπα, κάποτε και ο Τσέρτσιλ χρησιμοποιούμε μόνο τα στατιστικά, στοιχήματα, τα στατιστικά στοιχεία που εξυπηρετούν τα επιχείρημά μας αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο. Πάντως, ό,τι στοιχεία και να έχουμε για το κόστος, σίγουρα αυτό το τσίρκο με τα ταξίδια αυτά τα συχνά οικονομίες δεν πρόκειται να μας επιτρέψει σε ό,τι αφορά το αντιστάθμιση αποζημίωση που θα πρέπει να δοθεί στη Γαλλία θα πρέπει να δοθεί φυσικά κάτι. Αλλά αν έχουμε μερικές από τις συνόδους κορυφής ε, που από άψη κυκλοφοριακής συμφόρησης καλύτερα μην γίνονται στις Βεξέλλες, θα γίνονται στο Στρασβούργο. Έτσι θα έχουμε και προβολή του Στρασβούργου και όλα τα φώτα στραμμένα προς εκεί. Γιατί όχι λοιπόν. Και έτσι δεν θα γίνονται και δεν θα έχουμε τη μεταφορά του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά θα αναφέρεται στην ε, γραμματότηση. Περιμένουμε με ανυπομονησία λοιπόν να τη διαβάσουμε. Ίσως περιλάβετε και κάποια, κάποια συγκριτικά στοιχεία. 29 Αυγούστου λέει ο πρόεδρος η προθεσμία. Α, συγγνώμη, όχι. 16 Ιουλίου. 16 Ιουλίου μέχρι το μεσημέρι λέγει η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών ε, για να πάει στην αύξηση 17 του μηνός και στη δική μας επιτροπή στις 5. Αυτά, εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη, λύεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα να οργανώσω, θα ήθελα να είχα οργανώσει μια δεξίωση για να σας ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ιδιαίτερα τους εισηγητές για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τη γραμματεία, τους συνεργάτες, όλους όσους ε, εργάστηκαν τόσο σκληρά στις διαπραγματεύσεις αυτές τις δύσκολες και πολλές φορές εκνευριστικές. Πολύ θα ήθελα λοιπόν να μπορούσα να οργανώσω τέτοια δεξίωση, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Πάντως ευχαριστώ θερμά όλους όσους είναι παρόντες εδώ. Αναβάλλεται η δεξίζη για μετά τις θερινές διακοπές. Τότε θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα γιορτάσουμε τις προσπάθειες και τα επιτέγματά μας και θα ευχαριστήσουμε έτσι και εμπράκτος τους συνεργάτες μας για την αξιέπαινη τους προσπάθεια και το εξαιρετικό τους έργο. Μερικοί από εμά θα βρεθούμε στη Ουάσιγκτον. Δυστυχώ δεν θα συναντηθούμε με του συναδέλφου τη Επιτροπή ΕΚΟΝ, αλλά είμαι βέβαιο ότι και μεταξύ μα θα περάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, επικοδομητική και απολαυστική εβδομάδα στη Ουάσιγκτον. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρία.